παρατηρήσεις για τα πρακτικά και έτσι θεωρείται ότι κυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Κάποιες παρατηρήσεις για την έναξη της συνεδρίασης. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης. Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σήμερα στην Φλωρεντία και όπως γνωρίζετε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έχει την έδρα του στην Φλωρεντία και το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ η Γιορτή της Ευρώπης διεξάγεται εκεί Υπήρξε και μια συνεδρίαση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συναντήθηκα και με φοιτητές του Πανεπιστημίου. Είναι η 61η επέτειος της ε, διακήρυξης του Ρομπέρ Σουμάν διακήρυξη που οδήγησε μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. <clears throat> Πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα. Θα ήταν περήφανο ο Ρόμπερ Σούμαν για αυτά τα οποία πετύχαμε. Οι πατέρε οι ιδρυτέ γνώριζαν ότι οι κρίσει υπάρχουν για να τι ξεπερνάμε. Και ότι χρειαζόταν ένα καλύτερο μέλλον για την Ευρώπη, ώστε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο μέλλον για την Ευρώπη. Γι' αυτό προσβλέπουμε με ελπίδες ε, προς το μέλλον σε αυτή τη συγκυρία. Επόμενη πληροφορία που θα ήθελα να σας δώσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα είναι πλέον πλήρες μέλος της, Ευρω... της ε, παγκόσμιας κοινότητας, της παγκόσμιας κοινότητας. Στις 3 Μαΐου τα Ηνωμένα Έθνη δέχθηκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό αυτό το καθεστώς και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να προσφωνήσει και να απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι επίτευγμα κοινό της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε με μία φωνή ενωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντική η δράση και η δραστηριοποίηση με στένος σε αυτή τη συγκυρία γιατί είναι μια χρονική συγκυρία που πρέπει να δράσουμε όλοι μας και να δρούμε και στην Βόρεια Αφρική και στη Συρία και στον παχρένο όπου βλέπουμε κρίσεις να ξεδιπλώνονται μπροστά μας, ε, εξεγέρσεις. Στις 17 Μαΐου θα γιορτάσουμε την επέτειο κατά της ε, ομοφοβίας. Δυστυχώς παγκόσμια πρέπει να πούμε ότι διώκονται άνθρωποι και σκοτώνονται, δολοφονούνται ακόμα επειδή είναι ομοφιλόφιλοι. Στις συνθήκες και στην χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για να μπορέσει να ξεριζώσει, να εκριζώσει την ομοφοβία. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει, ούτως ή άλλως έχει καταδικάσει την θανατική ποινή που έχει επιβληθεί και επιβάλλεται σε άτομα από το, τις αρχές του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ της συμφιλίωσης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Και τώρα περνάμε στην κανονική μας εργασία σύμφωνα με την ημερησία διάταξη και πρέπει να πω ότι από πλευρά Ντε Παλέστρης εθίγει ένα θέμα υπήρξε ένα αίτημα το οποίο επαναληφθήκε του κ.